Good morning, dear colleagues. As uh, our chair, Mr. Cassini, announced yesterday that he had to fly back to Italy. Δυστυχώς ο πρόεδρος χρειάστηκε να φύγει χθες για Ιταλία, γι' αυτό θα προεδρεύσω εγώ λοιπόν. Σας καλημερίζω. Ανακοίνωση. Να για τις ε, διαδικασίες έγκρισης του προπολογισμού του 2014 η ομάδα μου αποφάσισε να ορίσει εισηγητή. Επίσης η κυρία Γκέραντ Χέφνερ πήρε μια έκθεση για την έκθεση της πρωτοβουλίας για τα θεσμικά οι τέσσερις εξής συστάθηκαν. Κασπόφσκι από το ΕΛΚ, Ρομπέρτο Γκαλτιέρη από εμά. Και για γνωμοδότηση της Επιτροπής ΝΟΜ, Γιούρι, η κυρία Αναγέτανάκη. Νάκη. Δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση για τον κανονισμό του προσωπικού και αν δεν ακουστούν αντιρρήσεις για όλα αυτά που σας λέω θα εγκριθούν αυτά που είπα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο. Με μεγάλη χαρά δίνω το λόγο στον κύριο Χέφνερ για να μας αναφέρει τη γνωμοδότησή του. Έχουμε λίγο χρόνο για αυτό το σημαντικότατο θέμα. Η Επιτροπή ΕΛΕΦ η αρμόδια για την ουσία και εμείς γνωμοδοτούμε. Ορίστε κύριε Χέφνερ μου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Τον επόμενο χρόνο, δηλαδή το 2013, θα είναι η χρονιά του πολίτη. Αυτό προέκυψε μετά από πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κατέθεσε ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, και Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Κομισιόν ε, για αυτή την πρόταση. Η εκπρόσωπος Κομισιόν, η κυρία Μπερνάρ, είναι, βρίσκεται εδώ για να σας εξηγήσει περαιτέρω αν θέλετε λεπτομέρειες για το σχέδιο αυτό. Το σχέδιο λοιπόν εστιάζεται σε θέματα των ελευθεριών του πολίτη, και κυρίως ε, σε όλο αυτό την προβληματική που ε, αναφέρεται ως ελευθερία κινήσεων, η κινητικότητα. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ε, ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Κατά την άποψή μου λοιπόν η πρόταση που γίνεται είναι πολύ καλή. Εμείς ε, δεν είμαστε η επί αρμόδια επιτροπή, είμαστε συμβουλευτική επιτροπή και τα θέματα τα οποία τίθενται εδώ νομίζω ότι θα στηθούν διεξοδικότερα σε άλλες ε, αρμόδιες επιτροπές, κυρίως στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Εμείς τώρα αυτό το οποίο ε, μπορούμε και πρέπει να εκφράσουμε στη γνωμοδότησή μας είναι το εξή. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Χρονιά των Πολιτών ε, μπορεί να αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένη. Συνολικά βρισκόμαστε σε δύσκολη περίοδο στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τους ε, μηχανισμούς αντιμετώπισης των κρίσεων και έχουμε τις πολιτικές ε, που επηρεάζονται από όλα αυτά. Σε πολλά κράτη-μέλη για τους πολίτες λαμβάνονται αποφάσεις ε, που συνεπάγονται ε, πολύ δυσάρεστες ε, συνέπειες αλλά οι πολίτες ε, δεν μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις αυτές και αυτή είναι η μεγαλύτερη μου ανησυχία όσον αφορά τη μελλοντική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή όλο και περισσότερο οι πολίτες ε, θα αισθάνονται ως ε, ουραγή, ως ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή την χρονιά των πολιτών οφείλουμε να την εκμεταλλευτούμε για να αποδιώξουν αυτό το συνέστημα. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσουμε όλα εκείνα τα οποία ξεπερνούν την ελευθερία του πολίτη και που έχουν σχέση με την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Αναφέρομαι κυρίως ε, στη συμμετοχή σε εκλογές, την ε, εκμετάλλευση συγκεκριμένων δικαιωμάτων, τη δυνατότητα συμμετοχής. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το εξής, να προχωρήσουμε μεθοδικά Δηλαδή όχι μονόπλευρα να ε, προβούμε σε ανακοινώσεις που απευθύνονται στον πολίτη, αλλά να αναζητήσουμε τρόπους για το πώς οι ίδιοι πολίτες μπορούν να υποβάλουν τις ε, ερωτήσεις τους ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ερωτήσεις που αφορούν στη συμμετοχή τη δική τους στην Ένωση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο στην προτινόμενη γνωμοδότηση εγώ καταθέτω κυρίως ε, προτάσεις οι οποίες ε, ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση που μόλις τώρα σας ε, περιέγραψα. Εγώ προτείνω Παραδείγματος χάρη να υπάρχει ένας Ευρωπαίος εντεταλμένος για τη συμμετοχή των πολιτών. Ένας εντεταλμένος ο οποίος θα έχει το καθήκον να καταγράφει τη συμμετοχή των πολιτών να αξιολογεί, να ελέγχει αυτή τη συμμετοχή και να ξεκινάει από προτάσεις που καταθέτουν οι ίδιοι πολίτες. Ε, πώς προτείνουν οι πολίτες ε, το δικό τους το ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιες θεωρούν ότι είναι οι δυνατότητές τους να εκφράζονται. Ο ρόλος αυτός πρέπει να ενισχυθεί. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να εκπέμψουμε ένα σημαντικό μήνυμα για το πώς είναι δυνατόν να λάβουμε σοβαρά τους πολίτες έτσι ώστε ο διάλογος με αυτούς να μην αντιμετωπίζεται ως ε, μια μονόπλευρη σχέση αλλά να αντιμετωπίζεται ως μια σχέση όπου εισακούεται η άποψη του πολίτη και κατόπιν τούτου οι προτάσεις ε, οι δικές μου ακολουθούν ε, αυτή την κατεύθυνση. Ένα άλλο θέμα το οποίο επιθυμώ να αναφέρω αφορά στη χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος με ένα εκατομμύριο μάρκα, λέει ο μιλητής, μάρκα. Κατά την άποψή μου, αυτό το ποσό δεν επαρκεί. Και κατόπιν τούτου ε, πρέπει να ε, εκταμιεύσουμε περισσότερα κονδύλια. Θα ήθελα λοιπόν ε, προς το παρόν τουλάχιστον να παραμείνω σε αυτά και αργότερα θα ήθελα να ακούσω και ποιες είναι οι δικές σας απόψεις Κατέθεσα λοιπόν για πρώτη φορά αυτή την πρόταση έτσι ώστε από τη συζήτηση να λάβω και εγώ ε, προτάσεις, ε, να ακούσω κριτική και στο τέλος ε, να μπορώ να καταθέσω μία πρόταση επί της οποίας θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Και στο τέλος της συζήτησης θα αναφέρω συγκεκριμένες προτάσεις. Thank you very much, dear colleague. να καλωσορίσω τον συνάδελφο που ήρθε σε, στη συνεδρίασή μας ως νέο μέλος. Ελπίζω να εξοικειωθείτε σύντομα. Ο Άντριου Ντάφ νομίζω ότι είναι αυτός που θα ήθελε τον λόγο. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν σχόλια να διατυπώσουν. Ωραία, σημειώνω. Βέβαια και εγώ. Επειδή είμαι σκιώδης θα λάβω το λόγο, αλλά πρώτα απ' όλα να ακούσω τους συναδέλφους. Τον Άντριου καταρχάς. Καλημέρα. Νομίζω ότι καλό θα ήταν πρώτα να ακούσουμε και την Κομισιόν. Ή τέλος πάντων στην ε, διάρκεια της συζήτησης να ακούσουμε την Κομισιόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτό το πρώτο σχέδιο γνωμοδότησης. Σε αυτό βέβαια δεν βλέπω πρόταση για τη δημιουργία ε, ενός νέου οργάνου, δηλαδή ενός ε, διαμεσολαβητή Ευρωπαίου για τα άνθρωπα δικαιώματα, αλλά ενστικτό να σας πω πώς αντιδρώ σε όλα αυτά εγώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση. Όπως κάνουμε γενικά με τη δημιουργία νέων ε, φορέων. Θελεστικών οργανισμών. Δεν θέλουμε να κάνουμε ιδιαίτερα πολύπλοκη την ευρωπαϊκή δομή. Γιατί αυτό θα προκαλέσει ακόμη περισσότερη σύγχυση από αυτή που ήδη δεν κατέχει τους πολίτες. Άρα αυτό το, Ευρωπαίο, το έτος των Ευρωπαίων πολιτών, το Ευρωπαϊκό έτος πολιτών πρέπει, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για αυτούς, να είναι μεγαλύτερη απλούστευση και διευκρίνηση αποσαφήνιση των δομών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να επιδιώξουμε. Επίσης πιστεύω ότι εάν μπορέσουμε φέτος ή στο έτος αυτό μάλλον να ολοκληρώσουμε και την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο ECHR, αν δηλαδή προσχωρήσουμε στη συνθήκη ως ένωση, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία. Υπάρχουν κάποια θέματα που εκκρεμούν ακόμη και είναι σημαντικά και ενδέχεται να καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο την ε, ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων τη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό. για να έχουμε επιτύχει μια κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ομοιόμορφη, καθολική. Και αυτό θα το πετύχουμε με την προσχώρηση στη συνθήκη για τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν ε, καταγγελίες των πολιτών parliamentary elections Θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν να τα αντιμετωπίζουμε άμεσα. Είτε μέσω του χάρτη, είτε μέσω των συνθήκων. ή μέσω της ε, σύμβασης. Inside, uh, Πρέπει να δείξουμε ότι ως Κοινοβούλιο αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην προσχώρησή μας σε αυτή τη σύμβαση. Στην ε, δε ε, αργή πρώτων διαπραγματεύσεων οφείλονται προβλήματα και αυτή την καθυστέρηση πρέπει να την επισημάνουμε. Έχουμε και τις ευρωεκλογέ και ιδίω το έτος πριν τις ευρωεκλογέ είναι ένα έτος που θα πρέπει άμεσα να δείξουμε στους πολίτες μας, στους ψηφοφόρους, τα ωφέλη που δεν είναι και τόσο προφανή για πολλούς πολίτες. And finally, can I congratulate Gerald on composing in his... Τέλος ένα ε, σχόλιο σε σχέση με την πρώτη τροπολογία. Μια πάρα πολύ μακρά, η πιο μακρά, ε, μακροσκελής πρόταση ε, στα αγγλικά τουλάχιστον δεν έχω δει πιο μακροσκελή ρεκόρ. Αυτό ήθελα να πω. Σας κατευχαριστώ για τα σχόλιά σας, κύριε Βορόντσε. Ευχαριστώ. Η ηθαγένεια της Ένωσης δεν μοιάζει με τις εθνικές ηθαγένειες. Βέβαια η Ένωση λέει ότι τάχα δεν είναι κράτος. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι αφού απαιτούμε η ευρωπαϊκή ηθαγένεια να συμβαδίζει με κάποια εθνική ηθαγένεια, μπορεί να μπερδευτούν τα πράγματα. Ας πούμε η βασίλισσα Ελισάβετ η δεύτερη είναι και πολίτης της Ένωσης θεωρείται μαζί με τη βασιλική της ιδιότητα. δεν λέμε ποτέ ποια είναι τα καθήκοντα του πολίτη, μόνο για τα δικαιώματα μιλάμε. Το 13 έμαθα ότι θα είναι έτος ευρωπαϊκής ηθαγενείας ή του Ευρωπαίου πολίτη. Μόλις το άκουσα αυτό, κόντεψα να πάθω τα μπλά, διότι αυτό μπορεί να σήμαινε ότι το 14, το 15 κλπ. δεν θα είναι του πολίτη κράτη. Ε, χρόνια. Οι εθνικές ηθαγένειες συνήθως καλύπτουν και την περίπτωση που κάποιος αρνείται την ηθαγένειά του ή του αφαιρείται. Αλλά η ευρωπαϊκή ηθαγένεια εφαρμόζεται με μια διαδικασία που ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο για τα συνδικάτα, δηλαδή όσο πληρώνουν. Δυστυχώς δεν προβλέπεται όμως κανένα έγγραφο έντυπο με το οποίο να κάνει κανείς αίτηση, γιατί πολλοί θα ήθελαν να αρνηθούν την ευρωπαϊκή τους ηθαγένεια και δεν μπορούν να το πράξουν. Είτε το έντυπο έχει κρυφτεί και δεν υπάρχει, είτε είναι στα υπόγεια της Κομισιόν κρυμμένο. Ευχαριστούμε πολύ. ναι. Χαίρετε. Το 13 είναι το έτος των πολιτών λένε. Στο έγγραφο του κυρίου Χέφνερ αναφέρεται η ελευθερία της μετακίνησης. Αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο τι βλέπουμε. Ότι δεν ελέγχονται πια τα υγειονομικά και έχει ξαναεμφανιστεί η φυματίωση. Ρουμανικές συμμορίες κλέβουν τα πάντα, ακόμη και μαστίχες. Ο κύριος Χέφνερ λέει ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι πολίτες. Ε, όντως αυτό καταλαβαίνουν, ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έρχονται τόσοι μετανάστες από τις άλλες ενωσιακές χώρες και καμιά φορά μιλούνται δέκα γλώσσες στο ίδιο σχολείο. Πώς θα αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς τους διαφορετικούς λαούς οι οποίοι επιμένουν αμέσω να παίρνουν δικαιώματα αλλά δεν αναφέρουν υποχρεώσεις. Εμείς στη Βρετανία βλέπουμε ότι μένουν ατιμόρυτα τα περισσότερα εγκλήματα. Ενώ ξοδεύονται εκατομμύρια για προπαγάνδα υπέρ της Ένωσης. ο Ραφαήλ. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω τον Κέρχαρντ για την πολύ καλή του έκθεση. Τι να συμφωνήσω με τον Άντριου πάντως. Αυτό για το μεσολαβητή Μόνιμο γραφείο για έναν ειδικό εκπρόσωπο των πολιτών, κάτι τέτοιο. Τροπολογία 18. Κοιτάξτε, κάποιες φορές νομίζω ότι αναζητούμε νέους φορείς, θέλουμε να εισαγάγουμε νέες ιδέες, έχουμε δει την Επιτροπή Άφετ και άλλες επιτροπές να διατυπώνουν νέες ιδέες κτλ. Κάποιες φορές όμως ε, όλα αυτά αποδεικνύονται απογοητευτικά γιατί στην πράξη δεν υλοποιούνται ή δεν γίνονται σωστά. Υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις αλλά δεν πρέπει να, να αποσπάσουμε την προσοχή των πολιτών από άλλες εξελίξεις. Έχουμε την πρόσφαση στο χάρτη, έχουμε την ε, πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Δύο καινοτομίε πολύ σημαντικές. Έχουμε κάνει δηλαδή ένα ποιοτικό άλμα στις σχέσεις μας με τους πολίτες και νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε ακριβώς σε αυτό. Σε αυτό το ποιοτικό άλμα. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η συνειδητοποίηση των δύο αυτών σημαντικών καινοτόμων θα πρέπει να τις ε, προβάλλουμε. Έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο σημαντικές καινοτομίες θα πρέπει να διαδοθούν, να ε, γίνουν πιο γνωστέ πολίτες. Αυτό το κάνετε με την εκθεσή σα. Επίση για την παιδεία, οι πρωτοβουλίες, όλες αυτές καλέ είναι. Αλλά Εάν θέλουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα, είναι σημαντικοί οι πολίτες γιατί είναι σημαντικές οι δύο καινοτομίες αυτές. Συμφωνώ τώρα με τον Άντριου σε ό,τι αφορά τη δημιουργία αυτού του γραφείου, του νέου γραφείου που θα μας ε, βγάλει από την πορεία που έχουμε ακολουθήσει με επιτυχία μέχρι τώρα, σε ό,τι αφορά δηλαδή και την προσχώρηση μας στο χάρτη. Τα άλλα θέματα που ήθελα να πω έχουν ήδη αναφερθεί από τους προλαλήσαντες, οπότε περιορίζομαι στο να σας συγχαρώ για την έκθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα χαιρόμαστε πολύ γιατί είναι εξαιρετική εκπρόσωπος της Κομισιόν που είναι εδώ. Θα την καλωσορίσω, αλλά ε, να πω και εγώ μερικά πράγματα. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν είναι τέλεια, κάθε άλλο. Βέβαια ελπίζω η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να επιφέρει σημαντικέ αλλαγέ με, τον εισηγητή, με την εισηγήτρια την κυρία Τιγόνη Παπαδοπούλη. Έχω συζητήσει. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γκέρχαρτ και είμαι πεπισμένη ότι η γνωμοδότηση τη ΑΦΚΟ βρίσκεται σε καλά χέρια. Ξεκολουθώ να πιστεύω ότι ο τίτλο του έτου, θα πρέπει να 2013 Ευρωπαϊκό Έτο Ιθαγένειας, όχι πολιτών, έτσι νομίζω συμφωνήσαμε πριν. Ήταν μια πολύ προσεκτική επιλογή από πλευρά Κομισιόν, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να υιοθετήσουμε εμεί αυτή την προσέγγιση, ιδίω ένα χρόνο πριν τι ευρωεκλογέ. Και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει να αλλάξει ο τίτλο, όπω είχαμε ζητήσει το 2010. Εν γέννη τώρα συμφωνώ με την προσέγγιση του Γκέρχαρτ που στόχο έχει να διευρύνει ε, το όλο ευρω του έτου αυτού. Πολύ σωστή προσέγγιση. Η ελευθερία μετακίνηση πολύ σημαντικό θέμα. Στηρίζω και το στόχο του άρθρου 2. Χαίρομαι που ο εισηγητής συμπεριλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο άρθρο 4, παράγραφος 4, λέγοντας ότι αυτό το έτος θα μπορούσε και πρέπει να χρησιμεύσει ως μια πλατφόρμα για τις ευρωεκλογές του 2014. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συμμετέχει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο έτος αυτό. Βέβαια βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα την άποψη της Κομισιόν για το Κοινοβούλιο και γι' αυτό χαίρομαι που ο Γκέρχαρντ είχε αυτή την προσέγγιση και επίσης για την έμφαση που δίνει στη νέα γενιά. εκατομμύρια νέοι είναι άνεργοι στην Ευρώπη, άρα ένας λόγος παραπάνω να τονίσουμε την νεολαία. Η νεολαία είναι ο πλούτο μα και πρέπει οι νέοι μα να εκτιμήσουν και αυτοί την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω και όλοι οι πολίτε. Έχω κάποιε απορίε σε σχέση με κάποια σημεία. Θα ήθελα ο Γκέρχαρτ να δώσει κάποιε παραπάνω λεπτομέρειε. Μιλήσατε για έναν εκπρόσωπο για του πολίτε. Καλό είναι αυτό ω ιδέα, αλλά πώ θα λειτουργήσει στην πράξη και με τι προπολογισμό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Θα ήθελα επίση να μου πείτε τι εννοείτε με αυτά τα βήματα συζήτηση πολιτών, civic fora και συζητήσει για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Πάντως η εκθεσή σας είναι πάρα πολύ καλή, αλλά να ακούσουμε και την Κομισιόν. Αφού βέβαια ε, και μετά θα ακούσουμε τις δικές σας, τα δικά σας συμπεράσματα. Η Κομισιόν λοιπόν πρώτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον ε, εισηγητή για το πρώτο αυτό σχέδιο γνωμοδότηση. Να ευχαριστήσουμε και τους βουλευτές για τα σχόλια που έκαναν πάνω στην πρόταση. Καλωσορίζουμε τις τροπολογίες που έχουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση του έτους του έτους των Ευρωπαίων πολιτών. Και να πω κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τον τίτλο του έτους. Σκοπός μας είναι το επίκεντρο να είναι στους πολίτες. Στους πολίτες και όχι στην ηθαγένεια στο άτομο δηλαδή. Θέλουμε να βάλουμε τον πολίτη στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής διαδικασίας. Σε ό,τι αφορά την νομική βάση κατανοούμε την Επιτροπή σας ε, και το ενδιαφέρον που δείχνει στο να συμπεριληφθεί συγκεκριμένα στην πρόταση το σύλλογο των δικαιωμάτων που έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και συγκεκριμένα το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε και το θέμα της Ιθαγένειας. Η αναφορά όμως στο άρθρο 20 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρώτο, στην πρώτη ιδεολογική σκέψη, ε, στο recital 1, καλύπτει νομίζω την ανησυχία σας. Δείχνει την επιθυμία της Κομισιόν να ενημερώνει τους πολίτες περισσότερο για αυτό το στο δικαίωμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις δραστηριότητες και εμείς θέλουμε να ακούσουμε τις ανησυχίες, τις ιδέες ε, των πολιτών και αυτό θα το πετύχουμε μέσω ε, της ε, δημόσιας διαβούλευσης για την έκθεση στα γέννης. Θα έχουμε διάφορες συνεδριάσεις ε, στις χώρες μέλη με τις αντιπροσωπείες μας που θα βοηθήσουν. Επίσης θα συνεργαστούμε με όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και συγκεκριμένα και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και με την κοινωνία των πολιτών για την προετοιμασία του έτους αλλά και με τους εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών. Το ίδιο είχαμε κάνει όταν προετοιμάζαμε το Ευρωπαϊκό Έντος Εθελοντισμού ή με τον δομημένο διάλογο. Συναντώμεθα πολύ συχνά με προσώπου τη κοινωνία των πολιτών για θέματα που αφορούν την ηθαγένεια, ούτω ή άλλω. Σε ό,τι αφορά τώρα τον προπολογισμό. Περιορισμένο το ποσό βέβαια και σε αυτό οφείλεται σε τρει λόγου. Πρώτα απ' όλα, περιορισμένοι πόροι για τη συγκεκριμένη θέση του προπολογισμού, άρα δεν μπορούσαμε να είχαμε πιο πολλά κονδύλια Επίσης, σε καιρό λιτότητας δεν θεωρήσαμε σκόπιμο να δώσουμε περισσότερα χρήματα για αυτές τις δραστηριότητες. Και τρίτον, δεν πρόκειται μόνο για το προπολογισμό, αλλά και για τη δημιουργία συνεργειών. Ο στόχος μας είναι να κινητοποιήσουμε στρατηγικούς εταίρους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κοινότητας των εμπλεκομένων φορέων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώστε να υλοποιήσουμε δράσεις κάτω από την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Έτους για τους Ευρωπαίους Πολίτες 2013. Όλοι όσοι μπορούν λοιπόν να, έχουν, να προσεγγίσουν τους πολίτες θα συμβάλλουν και έτσι θα έχουμε συμπληρωματικές πρωτοβουλίες που θα αναλυφθούν ε, δύο σπόρες από αυτούς τους οργανισμούς. Και εμείς βέβαια θα συμμετάσχουμε πλήρως. Και έχουμε και ε, μεγάλη έμφαση στην νεολαία, έχουμε την ε, νεολαία σε κίνηση και όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία θα αξιοποιήσουμε. Επίσης θέλω να τονίσω ότι δεδομένου του περιορισμένου χρονοδιαγράμματος που έχουμε στη διάθεσή μας για να διοργανώσουμε αυτό το έτος, στόχος μας είναι βέβαια να έχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση για να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατόν τις προπαρασκευές συνεργαζόμενοι με όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι το ευρωπαϊκό έτος είναι ένα μόνο εργαλείο μεταξύ πολλών άλλων. Άρα δεν μπορεί να έχει ως στόχο να υλοποιήσει πάρα πολλούς στόχους από πολλές πολιτικές. Και υπάρχουν και άλλα εργαλεία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι με το έτος αυτό να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση, να δώσουμε πλατφόρμα στους πολίτες για να ακουστεί η φωνή τους και ανησυχίες τους συνεχείς συζητήσει για την έννοια τη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Θα, και, θα βοηθήσουμε και στη διαδικασία για την εκπόνηση μελλοντική έκθεσης Ιθαγένειας και θα δούμε τι μέτρα θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε. Ελπίζουμε λοιπόν να έχουμε το το δυνατό συμφώνη για να μπορέσουμε και εμείς να αρχίσουμε τη συνεργασία μας με εσά και με άλλους ε, φορείς για να έχουμε ένα επιτυχημένο έτος. Πρόεδρος, μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτησή μου. Γιατί άλλαξε ο τίτλος. Και αντί να μιλάμε για Ευρωπαϊκό Έτος Φαγένες, μιλάμε για Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών. Είναι κάτι που δεν έχετε διευκρινίσει. Είπα στην αρχή της παρεμβασής μου ότι αλλάξαμε τον τίτλο γιατί θέλαμε να επικεντρωθούμε στον, στο άτομο ε, και όχι σε κάποια αρχή προτιμήσαμε να επικεντρωθούμε στον πολίτη και όχι στην ηθαγένεια. Η πρόεδρος είναι ένα μικρό σχόλιο όμως. Εμείς, οι ευρωβουλευτές, αλλά στο κοινοβούλιο, είμαστε φωνή του λαού, φωνή των πολιτών. αν αποφασίσαμε κάτι που το κάναμε για τη θεώρηση ότι είναι καλό για τους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί το αλλάζει τώρα η Κομισιόν. Η ευρωπαϊκή ηθαγένεια είναι μια ευρύτερη έννοια από την έννοια Ευρωπαίος πολίτης. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά, αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσω για όλους μας. Μήπως θα μπορούσατε να μας πάρετε πιο σοβαρά υπόψη. Γιατί ήταν απόφαση αυτή, δική μας, για, την αλλαγή ε, για, την, για τον τίτλο μάλλον. Νόμιζα ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε και να συνεννόμαστε καλύτερα. Το θέμα είναι σοβαρό. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε έτσι τους τίτλους, χρειάζεται διαβούλευση. Ε, αυτό θέλω να το θέσω υπόψη σας. Πάντως σας ευχαριστώ. Και τώρα ζητώ από τον εισηγητή μας να σχολιάσει και να απαντήσει τα ερωτήματα. Äh, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίως ε, ευχαριστώ πολύ τους ε, συναδέλφους ε, για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που είπαν και ευχαριστώ και την κυρία Μπερνάρ και την πρόεδρο. θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα που εφήγησαν. Πρώτον, όσον αφορά την επικεφαλίδα. Ε, και εγώ ε, το σκέφτηκα έτσι πολύ, με απασχόλησε πολύ και συμφωνώ με αυτό που είπε η Πρόεδρος. Όμως, ε, παρόλα αυτά, εγώ θα προτιμούσα Year of the Citizens και όχι of the Citizenship, δηλαδή η χρονιά των πολιτών και όχι της ηθαγένειας. Αυτό προτιμώ. Είναι καλύτερα να προβάλλουμε τους ε, μεμονωμένους ε, πολίτες, τους ανθρώπους και όχι τόσο την αρχή. Βεβαίως αυτό πρέπει να το κάνουμε με σοβαρότητα. Δηλαδή δεν θα πρέπει να πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο αναφέρεται έτσι σε αφηρημένες αρχές, να είναι ένα σχέδιο το οποίο λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον πολίτη και τον τοποθετεί στο κέντρο των διαδικασιών. Ε, μετά, αναφερθήκατε στο φόρουμ. Τι θα είναι αυτό το φόρουμ. Θα είναι ε, ένας ε, διαρθρωμένος διάλογος με τους πολίτες, με την κοινωνία των πολιτών. Να υπάρχει δηλαδή ένας ε, διάλογος για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Και έτσι να... Έχουμε και τον Ευρωπαίο Συντονιστή έναν ε, συντονιστή ο οποίος ε, θα ασχολείται με τον, ε, τον απασχολεί για το τι υπάρχει και ποια είναι τα προβλήματα. Και ίσως μπορούμε να επισημάνουμε και το εξής. Εν τω μεταξύ, σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχει συντονιστής και διαμεσολαβητής μάλλον. Και όπου υπάρχει, αυτό και πολύ σωστό. Αυτό που με απασχολεί είναι το εξής. Η συμμετοχή στη δημοκρατία, η ευρωπαϊκή ηθαγένεια, αυτά κατά κάποιον τρόπο ε, θεωρούνται αυτονόητα. Δηλαδή, τι σημαίνει, έχουμε υπουργεία για μονομένε εκδικευμένε πολιτικέ για την πολιτική μεταφορών, την πολιτική γεωργία, αλλά δεν έχουμε κανένα που να ασχολείται με τα προβλήματα των πολιτών όπως το τοποθετούμε εμείς, όχι δηλαδή με διαμαρτυρίες, εφέσεις και παράπονα, αυτά δηλαδή που κάνει ο διαμεσολαβητής, κάποιον άλλον που να ασχολείται με το πώς εμπλέκονται οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς ασκούν τα δικαιώματά τους και πώς μπορούμε να διευρύνουμε περαιτέρω τα δικαιώματα αυτά. Εγώ κάτι τέτοιο έχω κατά νου. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προηγουμένως ε, σας το είπα, σας το εξήγησα, γιατί θεωρώ ότι αυτό, αυτή η πρόταση είναι η πιο ε, προκλητική από τις άλλες ε, που κατέθεσα και εξάλλου αυτό φάνηκε και από τη συζήτηση που ακολούθησε. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ τους συναδέλφους αυτό που τώρα σας είπα να το ξανασκεφτείτε και στην επόμενη συνεδρίαση ε, θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε για την έκθεσή μου. Κατά τα άλλα, εσείς αναφερθήκατε πρόσβαση στην ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό ε, το βρίσκω σημαντικό. Ε, θα το συμπεριλάβω στην εκθεσή μου και θα το προβάλλω περισσότερο. Κατά τα άλλα, στις άλλες παρεμβάσεις δεν άκουσα από κάποιον να μου έκανε μια συγκεκριμένη πρόταση που να μπορώ να συμπεριλάβω στην εκθεσή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς και, λέει η Πρόεδρος, να σας ενημερώσω ότι η 6η Μαρτίου είναι η διορία για την ε, κατάθεση τροπολογιών. Και εάν ε, συμφωνείτε, ας πάμε στο επόμενο ε, σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ο συγητής ήρθε, τον καλωσορίζουμε και θα ήθελα να σας παρακαλέσω τα σημεία 5 και 6 να τα παρουσιάσετε ε, με μία και μόνο παρέμβαση, να τα συνδυάσετε. Φαντάζομαι όλοι θα συμφωνούν. Yeah. Share is okay. Uh, eu, eu uh, uma vez que se trata de um relatório uh, apresentado em português, vou usar a língua portuguesa. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω πορτογαλικά γιατί τα έχω μπροστά μου στα πορτογαλικά. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Μέντεφ Δεβίγο, τον πρώην συνάδελφο, που πλέον είναι Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων της Νέας Ισπανικής Κυβέρνησης. Διότι τον ευχαριστώ διότι ένα σημαντικό κομμάτι τη δουλειά το έχει ο ίδιο επιτελέσει. Ήδη είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις ε, στην Επιτροπή και γενικώ και οι επαφές που είχαμε βοήθησαν πάρα πολύ στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Πρόκειται για ένα σχέδιο απόφασης. για τη σύμβαση. Θα σας τα εξηγήσω όλα πάρα πολύ σύντομα. Δύο-τρεις ιδέες θέλω να εκθέσω. Πρώτα απ' όλα, το 2008 έγινε δημοψήφισμα για την ε, συνθήκη στην, ε, της Λισαβόνας στην Ιρλανδία με αποτέλεσμα ε, αρνητικό. Η Ιρλανδία εκλήθη να διατυπώσει μια θέση και μετά να διενεργήσει ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Τον Ιούλιο έγινε δεκτό, έγινε μια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας ζήτησε εγγύηση σε τρεις τομείς. Πρώτον, δικαίωμα στη ζωή, την οικογένεια και την εκπαίδευση. των χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και με κάποιες αρμοδές που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας φοβόταν η Ιρλανδία ότι ενδεχομένω ε, τεθούν σε κίνδυνο κάποιες διατάξεις ε, του συντάγματος της χώρας για τη ζωή, την οικογένεια και την εκπαίδευση, την παιδεία. Ένα αυτό. Δεύτερον, φορολογικό θέμα, είναι και πιο γνωστό. Η Ιρλανδία και ε, κυρίως για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, έχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς, ένα ιδιαίτερο σύστημα. Και έχει ένα σύστημα ενισχύσεων. Υπάρχει επίσης ε, η φορολόγηση των επιχειρήσεων, κατάφερε να το διατηρήσει η Ιρλανδία. Και υπάρχει και το καθεστώς ουδετερότητας, πολύ χαρακτηριστικό για την Ιρλανδία στα θέματα της ασφάλειας. Ζήτησε λοιπόν να έχει εγγυήσει για αυτά τα τρία θέματα όπως ε, προείπα η Ιρλανδία. Ασφάλεια, άμυνα, φορολογία επιχειρήσεων και ζωή, δικαίωμα στη ζωή, την οικογένεια και την παιδεία. Μετά από όλα αυτά, αυτό το οποίο εμείς έπρεπε να κάνουμε από εδώ και πέρα ήταν να καταλήξουμε σε δύο αποφάσεις. Καταρχάς να αποφασίσουμε κατά πόσον θα ανάγκαζαν όλες αυτές οι εγγύησεις ε, ε, να προχωρήσουμε σε μια τροποποίηση της συνθήκης ή σε ένα opting out, μια εξαίρεση. Και έπειτα να δούμε κατά πόσο εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπρεπε να ζητήσουμε να γίνει μία συνέλευση, convention, για να συζητήσει όλα αυτά. Μετά από σε βάθος ανάλυση όλων των ε, θεμάτων αυτών και προηγήθηκε μία ακρόαση πολύ σημαντική, ακούσαμε πάρα πολλούς, και με πολύ μεγάλη προσοχή και νομίζω ότι υπάρχει συνένεση ως προς τα ακόλουθα. Επί της ουσίας, οι εγγύησεις που ζητάει η Ιρλανδία δεν θέτουν να ε, στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ουσιαστικά εγγυώνται ότι η ερμηνεία της συνθήκης δεν θέτει σε κίνδυνο κάποια πολύ σημαντικά για την Ιρλανδία στοιχεία. Βέβαια αποχρώσεις υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι γενικά μπορούμε να πούμε ότι κανένα από τα τρία αυτά ζητήματα δεν δημιουργεί προβλήματα ή κάποιο κίνδυνο για την Ιρλανδία. Η Ιρλανδία ζητούσε κάποιες εγγύησεις. Σας έδωσα και τις εξηγήσει που ζητά η Ιρλανδία. Άρα, οι επιφυλάξει εντό εισαγωγικών, οι παρατηρήσει της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας που έγιναν αποδεκτές επί της ουσίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έγινε τελικά το δεύτερο δημοψήφισμα στις 2 Οκτωβρίου οι Ιρλανδοί τότε αποφάνθηκαν υπέρ τη συνθήκη Λισαβόνα ένα χρόνο μετά το πρώτο όχι που είχαν πει. Επαναλαμβάνω ότι αυτά τα τρία θέματα δεν ε, θέτουν ε, σε κίνδυνο σε καμία περίπτωση την ισορροπία τη συνθήκη Λισαβόνα. Για ερμηνείε πρόκειται ουσιαστικά. Σε ό,τι αφορά οικογένεια, εκπαίδευση και ζωή, ε, αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει και κάποια αρμοδιότητα εκεί, άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τώρα τη φορολογία, ναι, εκεί έγινε μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσον θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα εκεί. Στην έκθεση υπάρχει σχετική αιτιολογική σκέψη και θα πρέπει να προσθέσω το εξή. Έχει δείξει ιστορία ότι η στάση της Ιρλανδίας δεν εμπόδισε ε, τη χώρα να συμφωνήσει με τη διακυβερνητική συνθήκη. Οι διαδικασίες δηλαδή που έχουν να κάνουν με τον οικονομικό, φορολογικό, δημοσιονομικό συντονισμό έγιναν με συμμετοχή της Ιρλανδίας. Τι σημαίνει αυτό. Άρα και εδώ, στον τομέα της φορολογίας δηλαδή, λόγω της αυτής τριετούς εμπειρίας που έχουμε, μπορούμε να πούμε ότι μία εγγύηση ουσιαστικά ζητάει, δηλαδή και τίποτα παραπάνω. ουσιαστικά για την Ιρλανδία αυτό το οποίο ε, γίνεται είναι ότι διατηρείται το σύστημα φορολόγηση των εταιριών. Αν θέλετε τα μικρά γράμματα. Αυτό, αυτό είναι το όλο θέμα. Το βασικό θέμα. Και δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Έρχομαι στο τρίτο σκέλος που είναι άμυνα και ασφάλεια. Ούτε και αυτό το σκέλος μας δημιουργεί προβλήματα. Ναι, μεν είναι μακροσκέλο το κείμενο, αλλά το πνεύμα που διέπει αυτές τις προτάσεις ουσιαστικά ακολουθεί την κατεύθυνση που έχει οθετηθεί με τη συνθήκη σε σχέση με το πώς κάθε χώρα αποφασίζει να χειριστεί τα θέματα της ε, εκείνης πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, άρα είναι αποδεκτά τα όσα προτείνονται. Το σκέλος της ασφάλειας και της άμυνας δεν συζητήθηκε πάρα πολύ στην προκαταρκτική συζήτηση. Η υποχρέωση αλληλεγγύης, συνδρομής, σε μέλη που ενδεχομένως δεχθούν κάποια επίθεση. Η Ιρλανδία ουσιαστικά έχει αν θέλετε το μονοπόλιο ε, της απόφασης. Δεν ξέρω βέβαια μέχρι πού μπορούμε να, να φτάσουμε. Νομίζω ότι έχοντας μελετήσει πάρα πολύ καλά τα πράγματα, ε, μπορώ να πω ότι δεν εξαιρείται η Ιρλανδία, δεν αυτό εξαιρείται από την υποχρέωση αλληλεγγύης και συνδρομής. Έτσι τουλάχιστον ερμηνεύω εγώ. Δεν λέει όχι η Ιρλανδία, λέει ότι είναι στη διάθεση, είναι διατεθειμένη να ε, εφαρμόσει αυτή την ε, υποχρέωση, να εκτελέσει αυτή την υποχρέωση, αλλά θα επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα το πράξει. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Βέβαια να πω ότι στην προκαταρική συζήτηση δεν είχαν τεθεί έτσι τα πράγματα, αλλά... Για μένα ήταν το πιο λεπτό ζήτημα αυτό αλλά μετά από την ανάλυση που έκανα και κάνουμε γενικώ, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια που μα επιτρέπουν να δούμε ότι ούτε και εδώ ουσιαστικά απαιτείται κάποια τροποποίηση τη συνδίκη Λισαβόνα. Άρα, για να ε, συνοψίσω και να καταλήξω, θα περιμένω να ακούσω βέβαια και τις παρατηρήσεις των συναντέλφων, αλλά κατά τη δική μου άποψη, για κανένα από τα τρία θέματα τα οποία τίθεται δεν βλέπω να υπάρχουν προβλήματα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, δηλαδή ότι θα μπορούσε να ακυρωθεί, να παραβιαστεί, να πρέπει να τροποποιηθεί η συνθήκη, το αντίθετο. Και σωστά έκρινε την κατάσταση το Συμβούλιο. Η ερμηνεία που δινόταν σε κάποια άρθρα δεν έθετε υπό αφισβήτηση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι θέματα ερμηνεία, επαναλαμβάνω, για την Ιρλανδία. Και έπρεπε να δοθούν κάποιες εγγύησει. Αυτό ουσιαστικά είναι αυτό που κάνει το πρωτόκολλο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Άλλωστε, επαναλαμβάνω, πρόκειται για καθαρά ερμηνευτικά ζητήματα. Άρα, δεν νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και στην ε, σύγκληση μιας ε, συνέλευσης, convention. Εκεί καταλήγω εγώ. Έτσι ερμηνεύω εγώ τα πράγματα. Βέβαια, μπορεί κανείς να πάει πιο μακριά από αυτό που λέω εγώ στις δύο μου εκθέσεις. Δηλαδή να πει κανείς και δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι εμείς ως κοινοβούλιο θα έπρεπε να είχαμε μια πολιτική ευθύνη. Αν υπάρχει ένα κράτος που συμφώνησε με το Συμβούλιο πάνω σε μια συγκεκριμένη ερμηνεία της συνθήκης, Εμείς δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να παρέμβουμε για να, ε, γίνουν τελικά, ε, να γίνει μια επαναχώρηση, να γίνουν βήματα προς τα πίσω. Παναλαμβάνω, δεν δημιουργούν σημαντικά προβλήματα αυτά τα τρία θέματα. Εγώ έχοντας αναλύσει ε, τα ζητήματα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ήσυχοι. Εγώ προσωπικά έχω καθυσυχαστεί και νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας ώστε το πρωτόκολλο αυτό να ενταχθεί στο συνταγματικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εγγύηση για το ότι η ερμηνεία ε, των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγαίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Okay. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Δύο έχουν ζητήσει το λόγο. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιος άλλος που επιθυμεί να λάβει το λόγο. Ο κύριος Νταφ, παρακαλώ. Μάλιστα. Μια πρώτη, ένα πρώτο σχόλιο. Είμαι εισηγητής για ένα παράλληλο σχετικό θέμα και χθες οι συντονιστές είπαμε να ξανασυζητηθεί στην Επιτροπή um, we could not uh, reach a decision on the protocol. το πρωτόκολλο σε άλλη περίσταση. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τα δύο θέματα παράλληλα, το τσεχικό πρωτόκολλο και το Ιρλανδικό. Μπορεί βέβαια να καταλήξουμε σε αντίθετα συμπεράσματα, δεν ξέρω. Επίσης όμως νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα να μην συνδυάσουμε τα θέματα του τσεχικού ή Ιρλανδικού πρωτοκόλλου με την ένταξη της Κροατίας. Ξέρω ότι το Συμβούλιο αποφάσισε να κυρώσει τα τσεχικά και ιρλανδικά πρωτόκολλα ταυτόχρονα με την ένταξη της Κροατίας, αλλά και τότε και τώρα δεν θεωρώ ότι ήταν φρόνιμη αυτή η απόφαση του Συμβουλίου. Θα ήταν κρίμα η ένταξη της Κροατίας να επηρεαστεί αρνητικά από περιπλοκές ή καθυστερήσεις που οφείλονται στο Ιρλανδικό και Τσεχικό πρωτόκολλα. Στην παράγραφο 2 λοιπόν της έκθεσης πρέπει να αναφερθούμε στην... δεν πρέπει να αναφερθούμε καθόλου στο θέμα της νέας κυβέρνησης της Κροατίας. Τώρα επί της ουσίας. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Και δεν πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να ερμηνεύσουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας με τρόπο που να ξεπερνάει αυτά που προβλέπει. Το Κοινοβούλιο πρέπει να ασκήσει όση πίεση μπορεί επί των συναδέλφων μας του Συμβουλίου για να γίνει σωστή διαπραγμάτευση και να υπογραφτεί μια συνθήκη που να περιορίζεται σε αυτά που προβλέπουν οι συνθήκες. Βέβαια από πολιτικό ρεαλισμό καταλαβαίνω ότι μερικές φορές πρέπει κανείς να συνδυάζει και να συγκολλάει κατά κάποιον τρόπο και πρόσθετα πρωτόκολλα στη για να μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά δεν μου αρέσει αυτό. Και δεν πιστεύω ότι πρέπει να δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι θέλουμε κάτι τέτοιο. Συμμερίζομαι τις αμφιβολίες του Ραγκάλ σχετικά με την πολιτική ασφαλείας και άμυνας, ή τη μάλλον ασφαλείας και άμυνας στο πρωτόκολλο. Νομίζω ότι καθορίζει έτσι μια Ιρλανδική εξαίρεση στη συνθήκη της Λισαβόνας ως προς τα θέματα ασφαλείας και άμυνας και πρέπει να ξέρουμε τι λέμε όταν λέμε τέτοια πράγματα, τι εννοούμε. Επίσης νομίζω ότι στο άρθρο 2 για τη φορολόγηση ότι δεν ισχύει ότι δεν αλλάζει τίποτα η συνθήκη της Λισαβόνας για οποιαδήποτε χώρα μέλος. ως προς τις δικαιοδοσίες της Ένωσης για θέματα φορολογικά. Αν οι Ιρλανδοί το ερμηνεύουν έτσι, δικαίωμά τους. Αλλά εγώ δεν εγκρίνω, δεν εγκρίνω, δεν εγκρίνω αυτή την ερμηνεία. της φορολογικής πολιτικής, των ρητρών φορολογικής πολιτικής της Λισαβόνας. Πράγματι, μάλιστα θα έλεγα ότι τα γεγονότα μου δίνουν δίκιο. Ο κύριος Ραγκάλ δικαίωσα είπε ότι το σύμφωνο, το φορολογικό σύμφωνο έχει επηρεάσει άμεσα τις δικαιοδοσίες της Ένωσης ως προς τη φορολογική πολιτική. Και αναρωτιέται κανείς πώς θα μπορούσε ένα δικαστήριο να τετραγωνίσει αυτά τα πράγματα. Το άρθρο 2 λοιπόν του Ιρλανδικού Πρωτοκόλου πώς θα συνδυαστεί με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η Ιρλανδική κυβέρνηση δηλώνει ότι το πρωτόκολλο αυτό είναι πολιτικά σημαντικό για εκείνην. Αλλά για μας απλώς τεχνικό θέμα. Αυτό δεν το δέχομαι. Αν κάτι είναι πολιτικά σημαντικό για την Ιρλανδική κυβέρνηση, τότε είναι πολιτικά σημαντικό και για όλους τους άλλους. Ζητώ λοιπόν στην επόμενη μας συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή μας να ζητήσουμε από έναν εκπρόσωπο της Ιρλανδικής Κυβέρνησης να προσέλθει εδώ για να ανταλλάξουμε απόψεις επί της ουσίας ή της σημασίας του πρωτοκόλλου αυτού. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Φαίνεται λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, παραπλάνησε τους Ιρλανδούς για να εξασφαλίσει τον έτους ε, στο δεύτερο ε, δημοψήφισμα. Να δούμε τι θα γίνει με τους ε, Κροάτες. Τώρα λοιπόν ισχυρίζεται ότι αυτές οι διαβεβαιώσεις είναι νομικά δεσμευτικές και γι' αυτό λένε ότι δεν είναι απαραίτητο να συγκληθεί συνδιάσκεψη ε, με βάση το άρθρο 48 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά τα έχουμε ξανακούσει κατά το παρελθόν και όπως είπε και ο κύριος Νταφ στη δική του την παρέμβαση η ε, Βρετανική κυβέρνηση και η Τσεχική κυβέρνηση έδωσαν τη ε, ότι ο χάρτης ε, θεμελιδών δικαιωμάτων το λέω πολύ προσεκτικά, δεν τους αφορούν πλήρως. Το άρθρο 1, υποπαράγραφος 1 του πρωτοκόλου Αναφέρει μάλιστα ότι αποκλείονται ε, τα δικαστήρια, τα αρμόδια στην Πολωνία και στις εν λόγω χώρες να καταλήξουν σε ενέργειες ε, οι οποίες είναι ασύμβατες με το χάρτη. Και όπως ε, είπε και ο κύριος Ντάφ πριν από λίγες εβδομάδες, τώρα λοιπόν γνωρίζουμε από την περίπτωση C411 που αφορά έναν Αφγανό πολίτη ότι οι διαβεβαιώσεις του πρωτοκόλλου ήταν άχρηστες. Φαίνεται λοιπόν τώρα πλέον ότι η απάντηση στο να υπάρχουν άχρηστα πρωτόκολλα είναι το να μην επισυνάπτονται καθόλου τα πρωτόκολλα. Δηλαδή αν διαπιστώσει κανείς ότι αντιμετωπίζει ε, δυσκολίες λέγοντας ψέματα δεν λέει κανείς τίποτα. Η προθυμία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, να προβαίνουν σε άχρηστες διαβεβαιώσεις. Αυτό μας ε, θυμίζει έναν παλαιό, παλαιότερους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ε, οι οποίοι το 1938 είπαν για τον Τσάμπλιν ότι ήθελε κάποιον αυτόγραφο και το έδωσε. Αν θέλουμε λοιπόν τις ε, υπογραφές... Θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι η ε, συνθήκη της Λισαβόνας υπογράφηκε με ψεύτικες ε, υπογραφές. Έχει χαθεί όμως η ηθική διάσταση του όλου θέματος. Βεβαίως, η Ιρλανδική κυβέρνηση είναι είτε αφελής, είτε και ίδια ανηλικρινής, γιατί σε τελική ανάλυση δεν υπάρχουν τομείς ε, οι οποίοι ε, θα παραμένουν άθικτοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι όλη το σύνολο της νομοθεσίας ε, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπόκειται στην νομοθεσία που εκπονείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλοι δύο συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο ο κύριος ε, Χέφνερ και μετά ο κύριος ε, Μοράιρα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω να πω ότι συμφωνώ με αυτά που είπε ο και πιστεύω ότι αυτή την περίπτωση πρέπει να τη διαχωρίσουμε από ε, το πρωτόκολλο της ε, Τσεχικής Δημοκρατίας. Γιατί τα δύο πράγματα είναι παντελώς ασύνδετα μεταξύ τους. Και αυτό αφορά όχι μόνο στο περιεχόμενο, αλλά αφορά και στην προϊστορία και στη διαδικασία. Κατά την άποψή μου είναι τελείως διαφορετικό το κατά πόσον μετά από ένα δημοψήφισμα ακολουθούν συζητήσεις ε, σχετικά με κάποιες διαβεβαιώσεις που εδόθηκαν ως προς την ερμηνεία μεμονωμένων άρθρων για να επιτευχθεί η ε, συνένεση, η σύμφωνη γνώμη ε, σε μία συμφωνία και ως εκ τούτου η παραμονή μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελείως διαφορετικό αυτό από το να ε, λαμβάνεται μία απόφαση του Κοινοβουλίου η οποία απαιτεί εξαιρέσεις. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και όπως και στην περίπτωση της Τσεχίας, εδώ δεν τίθεται ε, θέμα για το σύνολο του Ευρωπαϊκού Χάρτη ή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, αλλά πρόκειται για την ερμηνεία μεμονωμένων διατάξεων. Αυτή ήταν η μία μου παρατήρηση και άλλη αφορά την ουσία, το περιεχόμενο, την ε, ερμηνεία όσον αφορά το δικαίωμα ζωής, το δικαίωμα οικογένειας, παιδείας, όπως και ο εισηγητής, θεωρώ ότι σε τελική ανάλυση όλα αυτά δεν είναι και τόσο τεράστια σημασία, γιατί έτσι κι αλλιώ και από τη σύμβαση δεν ρυθμίζει τίποτα το σπουδαίο. Λιγάκι διαφορετικά βλέπω το θέμα ε, στην πολιτική ασφάλειας, γιατί απλά διαρωτώ τι ακριβώς ε, εννοούμε στην πράξη με την ρήτρα ασφαλείας όταν υπάρχουν επιφυλάξεις. Συμφωνώ βέβαια με αυτό που ο κύριος ε, Πολ Ρέγγενς, ότι τουλάχιστον ε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες υποχρεώσει από τις οποίες να επιθυμεί να αποσυρθεί η Ιρλανδία. Και θα το παρακολουθήσουμε και θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Τώρα, έχω επίσης ε, πρόβλημα επί της ουσίας με την διαβέωση που δόθηκε για τη φορολογική πολιτική. Πρέπει όμως ε, να σας πω ότι εδώ δεν έχω τόσο μεγάλο πρόβλημα με το πρωτόκολλο, γιατί και με αυτό το πρωτόκολλο δεν ρυθμίζεται άμεσα κάτι που να αφορά στη συνθήκη της ε, Λισαβόνας και αυτά που ρυθμίζονται είναι εκτός των συνθήκων. Νομίζω όμως ότι μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταλήξουμε σε μία συζήτηση έτσι ώστε η αλληλεγγύη και η ανάληψη ευθυνών για τα δημοσιονομικά προβλήματα ορισμένων κρατών. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο και εάν υπάρχει ε, κάποια ελάχιστη αλληλεγγύη ως προς την φορολόγηση. Η Ιρλανδία, παραδείγματος χάρη, έχει ένα πολύ μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα και δεν διαθέτει επαρκή πόρους ε, για να καλύψει τις δαπάνες του κράτους. Παράλληλα όμως η Ιρλανδία έχει έναν από τους ε, χαμηλότερους, επιχειρηματικ... χαμηλότερους επιχειρηματικούς ε, στην Ευρώπη. Αυτό μακροπρόθεσμα δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου πολλά ρυθμίζονται από κοινού, καταλαβαίνετε αυτό απαιτεί να υπάρχει αλληλεγγύη. Γιατί σε τελική ανάλυση αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, μία χώρα ε, παίρνει περισσότερα από αυτά που δίνει. Και σε μία ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, κυρίως όσον αφορά την επιχείρηση, την φορολόγηση των επιχειρήσεων, είναι προφανές ότι θα πρέπει να προκύψει μεγαλύτερη κοινωτική αλληλεγγύη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, την παρατήρηση αυτή την κάνω παίρνοντας αφορμή από το πρωτόκολλο αυτό το οποίο συζητάμε όσον αφορά ε, στην αξιολόγηση, τη γενικότερη αξιολόγηση του συγητή, συμφωνώ επ' αυτής, μόνο που θεωρώ ότι εδώ στην περίπτωση δική μας ε, ε, δεν πρέπει να εκφράσουμε αντιλήσεις, σε αντίθεση βέβαια με το πρωτόκολλο της Τσεχίας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μορέρη είναι ο τελευταίος ομιλητής. Thank you. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα σας κάνω τα εξής σχόλια. Δύο τελείες. Καταρχάς, διαμαρτύρομαι εντόνως σχετικά με την ιδέα ότι παράτυπα έγινε η διαπραγμάτευση της συνθήκης της Λισαβόνας. Συζητήθηκε πολλές φορές και εγκρίθηκε πολύ νόμιμα. Από... Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει λοιπόν. Κανείς. Ούτε μπορεί να δεχθεί κανείς σιωπηρά και διαμαρτύρητα να ακούγονται τέτοιες κατηγορίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο ομόφωνα δεσμεύτηκαν ότι θα διευκρινίσουν κάποιες διατάξεις της συνθήκης προκειμένου να διευκολύνουν στην Ιρλανδία διαφορετική έκβαση του δημοψηφίσματος. Υπήρξε πολιτική ειλικρίνεια, πιστεύω, και τιμιότητα. Πρέπει λοιπόν να τηρηθεί και η υπόσχεση που δόθηκε. Αυτό ακριβώς που θέλουμε είναι η συμβιβαστική αυτή πρόταση στο Συμβούλιο να περάσει και να υλοποιηθεί. Σε ό,τι αφορά την Ιρλανδία δεν έχω καμία αμφιβολία προσωπικά. Δηλαδή κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει, κατά την άποψή μου. Άρα, που έχει η δική μου αμφιβολία, όπως λέει και ο Παόλο Ραζέλ, εδώ έχουμε να κάνουμε με πραγματικό opting out ή απλά είναι ερμηνευτικό το θέμα. Γιατί τα δύο πράγματα δεν είναι ταυτόσιμα, ούτε θα είχαν τις ίδιες επιπτώσεις. Εάν δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για μια απλή ερμηνεία της συνθήκης, και κατά το τρίτο σκέλος περιοριστικά, ε, περιοριστική ερμηνεία, Άρα η ερμηνεία του πρωτοκόλου είναι η αυθεντική ερμηνεία της συνθήκη, αλλά αυτό, προσοχή, δεν ισχύει μόνο για την Ιρλανδία, θα μπορούσαν και άλλες χώρες δηλαδή από τώρα και στο εξή να χρησιμοποιήσουν αυτή την ερμηνεία. Τώρα, αν μιλάμε για opting out της Ιρλανδίας, για εξαίρεση της Ιρλανδίας, αυτό αφορά μόνο και μόνο την Ιρλανδία. Τι προτιμώ εγώ αν με ρωτήσετε τώρα. Προτιμώ το δεύτερο, έτσι. Γιατί αυτή η ερμηνεία τουλάχιστον τι κάνει, διατηρεί ουσιαστικά την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για μία και μάλιστα περιοριστική ερμηνεία, απλά και μόνο. επηρεάζεται η εθνική πολιτική ασφάλειας και άμυνας με την κοινοτική πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι επηρεάζεται. Όποιο κράτος δηλαδή αντιμετωπίσει μια τρομοκρατική ή άλλη επίθεση υποτίθεται ότι πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη και συνδρομή από τα άλλα κρατημέλη. Αυτό δεν είναι το ίδιο με το να μπορεί να επιλέγει το κάθε κράτος πώς θα υλοποιήσει αυτή την αλληλεγγύη ή συνδρομή. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό το πρωτόκολλο είναι opting out της Ιρλανδίας ό,τι αφορά την πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Τώρα έρχομαι στο θέμα της φορολογίας. Ούτε και αυτό πρέπει να το εκλάβουμε ως μια απλή ερμηνεία, που είναι και πάρα πολύ περιοριστική μάλιστα. Ουσιαστικά είναι σαν να βγάζουμε το, τη σάρκα από τα οστά. Αυτό κάνουμε. Αυτό που πρέπει να αναγνωριστεί τελικά είναι ότι η Ιρλανδία βρίσκεται σε μια διαφορετική θέση. Ξεχωρίζει τη θέση από του άλλου 26. τη συνθήκη την ψηφίσαμε. Το θέμα είναι τώρα να την ερμηνεύσουμε. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση τη Ιρλανδία, το πρωτόκολλο εγώ το αντιλαμβάνομαι ω εξαίρεση τη Ιρλανδία και όχι ω ερμηνεία τη συνθήκη. γιατί αυτό θα μπορούσε, επαναλαμβάνω, να ισχύει για όλα τα άλλα κράτη-μέλη. Ο κ. Ρανζέλ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα σε ευχαριστώ. Για όσα είπατε όλοι. Βέβαια, ακολουθώ τη στάση του συναδέλφου Βιτάλ Μορέα. Αυτά που είπε δηλαδή για το όραμα του συναδέλφου Μπρόμς. Δεν το αφισβητώ αυτό. Για μένα είναι σαφές ότι δεν υπήρξε παρατυπία. Αντίθετα όλα γίνανε διαφανώς. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αν και συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο Χέφνερ, Of what? Δεν χρησιμοποίησα ως υπόδειγμα ή παράδειγμα την Τσεχία, γιατί Διαφωνώ με τον συνάδελφο Νταφ μόνο ως προς το εξής. Αν γίνει εξαίρεση για μία χώρα, τότε πρέπει κάθε χώρα να τη δούμε μεμονωμένα. Είναι θέμα σεβασμού στοιχειώδους. Κάθε χώρα που είναι μέλος της Ένωσης πρέπει να γίνεται σεβαστή πλήρως και δεν πρέπει λοιπόν τη θέση δύο, τριών, τεσσάρων χωρών να τη θεωρούμε ενιαία ή να της επιβάλλουμε μια λύση γιατί έχουμε πρόβλημα με κάποια άλλη χώρα. Δεν πρέπει να έχει πρόβλημα μια χώρα επειδή έχει δυσκολία μια άλλη χώρα. Πρέπει και τις 27 χώρες να τις σεβόμαστε την εθνική τους κυριαρχία και κάθε πρόβλημα να το λύνουμε μεμονωμένα. Και αυτό δεν μίλησα για την Τσεχία. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική από τις άλλες και κάθε χώρα πρέπει να την χάνει σεβασμού και με μονομένης ανάλυσης του Κενοβουλίου. Δεύτερον, από ό,τι βλέπω εδώ, ο συνάδελφος Μπρόγκς Έχει μία σφαιρική πολιτική θέση που τη σέβομαι αν και διαφωνώ. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα. Αλλά και ο Νταφ και ο Μορέρα έχουν ορισμένες αμφιβολίες ως προς την πολιτική ασφαλείας και άμυνας ή τουλάχιστον τη σχετική δήλωση. θα δεχτώ, θα παραδεχτώ τις αντιρρήσεις του κυρίου Μορέιρα γιατί είναι πιο πρόσφατες, τις έχω πιο πρόσφατες στη μνήμη μου. Όταν λέμε ότι η κοινή πολιτική δεν επηρεάζει θέματα ασφαλείας και άμυνας για κάθε χώρα μέλος, αυτό το λέμε και στο 42, δεύτερο εδάφιο διότι είναι σαφές ότι πράγματι δεν μιλάμε για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κάθε χώρας ως την πολιτική ασφαλείας και αμήνης. Αν μερικές χώρες είναι στο ΝΑΤΟ και θέλουν να παραμείνουν, τότε πρέπει να σεβαστούμε και τις άλλες που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Ακόμη λοιπόν και αν ορισμένοι έχουν την ερμηνεία α, υπάρχει και το γράμμα του σημείου αυτού που είναι σαφές. Δεν επηρεάζεται καμία ιδιαιτερότητα από καμία χώρα, σε καμία χώρα από το θέμα αυτό. Αυτά λέει το 42.2. Και ακόμη και στην περίπτωση υποχρέωσης βοήθειας δεν ξέρω πώς ακριβώς το λένε στα αγγλικά γιατί εδώ μπροστά μου το έχω στα πορτουγαλικά, ή η για να το πω έτσι. Είναι σαφές στο 42.7 ότι στην τελευταία φράση της πρώτης παραγράφου του 42.7 ότι δεν επηρεάζεται η ιδιαιτερότητα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας μερικών χωρών μελών. Εδώ το λέει, στη συνθήκη της Λισαβόνας το λέει. Δεν είναι τίποτα καινούριο. Θα θέλαμε ίσως να έχουμε μόνο την πρώτη φράση, αλλά υπάρχει και η δεύτερη. Και το μόνο που κυβέρνηση και ο Ιρλανδικός λαός ζήτησαν ήταν να θυμηθούμε ότι υπάρχει και η δεύτερη φράση, τίποτε παραπάνω. Βεβαίως πρόκειται για ερμηνεία, ναι, αλλά είναι θεμητή ερμηνεία και όχι και τόσο στενή. Το λέει εδώ, το λέει. Θέλω λοιπόν να πω ότι και για μένα όταν μελετούσα αυτή την περίπτωση είχα μια αμφιβολία ως προς την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, όχι για τη φορολογία, αλλά μετά όταν μελέτησα πιο συγκεκριμένα, πιο λεπτομερώς την κάθε φράση, κατάλαβα στο κείμενο της συνθήκης Λισαβόνας υπάρχει, δίνεται βάση για να υποστηρίξουμε την ερμηνεία ότι η Ιρλανδική κυβέρνηση, της Ιρλανδικής κυβέρνησης ή την ερμηνεία που θέλει να δώσει η Ιρλανδική κυβέρνηση. Τέλεια. Τέλος, Θα ήθελα να πω ότι για μένα είναι πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο να δεχτώ ότι πρόκειται εδώ για εξαίρεση και opting out. διότι υπάρχει και η θέση της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Και δεν υπάρχει χώρος εδώ για να δεχτούμε opting out μετά την κατάληξη, μετά την κύρωση της συνθήκης. Πολύ δύσκολο. Το πρωτόκολλο, το πνεύμα του πρωτοκόλλου δεν είναι αυτό που λέτε. Δεν είναι αυτό. Απλώς εδώ διασαφίζουμε τα πράγματα, αποσαφηνίζουμε. Νομίζω ότι σας έχω δείξει ότι δεν υπάρχει θέμα η τα σχόλια της Ιρλανδικής κυβέρνησης να είναι καινοτομίε. Όχι, αφού υπάρχει γραπτό στην τελευταία φράση του 47.2 και στην τελευταία φράση της πρώτης παραγράφου του 42.7. Υπάρχουν αυτά γραμμένα. Και αφού υπάρχουν γραμμένα πρέπει να τα σεβαστούμε και την ερμηνεία αυτών δεν πρέπει να τα θεωρήσουμε εξαίρεση και opting out. Πώς μπορεί να υπάρχει opting out όταν λέγεται ρητά στο κείμενο ότι θα σεβαστούμε την ιδιαιτερότητα της πολιτικής κάθε χώρας στα θέματα κοινή άμυνας και ασφάλειας. Νομίζω αρκούν αυτά. Αλλά να. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ καλά πηγαίνουμε προς τον χρόνο. Αλλά ο Άντριου, νομίζω για ένα λεπτό θα, θα ήθελε το λόγο. Ναι, ακούστε, νομίζω ότι μπαίνουμε σε δύσκολα χωράφια. Πολύ λεπτή η συζήτηση αυτή. Το άρθρο 42.2, δεύτερη υποπαράγραφος, νομίζω ότι καθιστά ξεκάθαρο το ότι υποχρεώσεις ορισμένων κρατών που είναι στο ΝΑΤΟ θα γίνουν σεβαστές που είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτό λέει. Το πρωτόκολλο δεν το λέει αυτό. Όχι και δεν το λέει, είναι ξαφές. Ρητός δεν το φαίνεται ότι δεν το λέει. Οι Ιρλανδοί βέβαια δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν θέματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω συζήτηση. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να επαναλάβω το αίτημά μου. Στην επόμενη συζήτηση του θέματος αυτού, δηλαδή 19 και 20 Μαρτίου, να παρακαλέσουμε να παρίσταται ένας εκπρόσωπος της Ιρλανδικής Κυβέρνησης. Να δώσω τώρα στον κύριο Ρανζέλη. Ναι. Για να δούμε. Θέλω να σας επενθυμίσω την πρώτη ε, πρόταση της Δευτέρας που μιλάω ότι θα επηρεαστεί ο ειδικό χαρακτήρα ε, τη πολιτική ασφάλεια και άμυνα ορισμένων κρατών. Και αυτό είναι που καλύπτει τελικά το Ιρλανδικό παράδειγμα. Μετά έχουμε τη δεύτερη πρόταση που μιλάει για το ΝΑΤΟ. Αλλά στην πρώτη πρόταση, σαφώς, γίνεται λόγος στη, για την ιδιαιτερότητα, των ιδιαίτερο χαρακτήρα τη εθνική πολιτικής άμυνα και ασφάλεια. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Γιατί γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει μόνο η Ιρλανδία που έχει μια ειδική αμυντική πολιτική. Έχουμε τουλάχιστον άλλε δύο, Αυστρία και Σουηδία. Όταν λοιπόν συντάχθηκε αυτό το κείμενο, ε, αυτοί που το συνέταξαν δεν σκέφτονταν μόνο την Ιρλανδία και έκλειναν τα μάτια του σε άλλε χώρε. Σκέφτονταν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και τα κράτη που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, ουδέτερα. Ε, μη ουδέτερ και τα λοιπά, δέσμευτη και μη. Λοιπόν, η πρώτη πρόταση της δεύτερης παραγράφου δεν μιλάει για τον ΝΑΤΟ, αλλά για την ιδιαιτερότητα του κάθε κράτους. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Είναι ξεκάθαρο. Δεν νομίζω λοιπόν Δεν νομίζω λέγω. Ότι χρειάζεται να έρθει εδώ η Ιρλανδική κυβέρνηση. Δεν υπάρχει τίποτα τόσο βαθύ που πρέπει να εξηγήσουν. Μην αναγάγουμε αυτό το θέμα σε πολιτικό πρόβλημα. Μην τα περιπλέξουμε τα πράγματα. Για να σας πω ακόμη και κάτι άλλο. Κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι εάν είναι κάποιο που πρέπει να εξηγήσει κάτι, αυτό δεν είναι η Ιρλανδική κυβέρνηση, αλλά είναι το Συμβούλιο. Άρα, δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια άμεση επαφή εδώ με την Ιρλανδική κυβέρνηση, γιατί το Συμβούλιο ήταν αυτό που δέχτηκε τη θέση τη ε, Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Αν λοιπόν έχουμε οποιαδήποτε αμφιβολία, ας θέσουμε το ζήτημα στο Συμβούλιο. θα πρέπει να πει το Συμβούλιο κατά πόσον πρέπει να συγκληθεί μια ε, συνέλευση, μια διάσκεψη διακυβερνητική. Οι σχέσεις που έχουμε εμείς είναι με το Συμβούλιο. Εκεί πρέπει να απευθυνθούμε, όχι προς την Ιρλανδική κυβέρνηση. Δεν θα ήταν ε, ε πρέπον και θα δημιουργούσε και ζητήματα συνταγματικού χαρακτήρα. Να οργανώσουμε ένα είδος ακρόασης της Ιρλανδικής κυβέρνησης στην Επιτροπή μας. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση Θα θεωρούσα ότι μπορούμε να πάμε πολύ γρήγορα σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος, ωραία. Άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις ψηφοφορίες. Νομίζω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε την σύσταση του εισηγητή που λέει ότι πρέπει να πάμε γρήγορα από εδώ και πέρα. Άρα θα έλεγα να ορίσουμε ως προθεσμία κατάθεση τροπολογιών την 6η Μαρτίου για να τηρήσουμε έτσι το ε, χρονοδιάγραμμα της ψηφοφορίας μας ε, στην ε, Επιτροπή και να πάει η έκθεση τον Απρίλιο στην Ολομέλεια. Αν βέβαια έχετε σχόλια, οι συνάδελφοι μπορείτε να καταθέσετε προπολογίες, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτό που είπε ο εισηγητής και να ορίσουμε την προθεσμία μας για τις 6 Μαρτίου. Να καλωσορίσω τον κύριο Ντομένιξη που αντικαθιστά τον κύριο Γκουαλτιέρη από τους σοσιαλιστές εδώ και να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες μας. Πρώτη έκθεση, ο Αλέν Λαμασούρ είναι εδώ, τον καλωσορίζω, είναι ο εισηγητής της πρώτης έκθεσης, ήμουν σκιώδης εγώ. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Προπολογία 1 του εισηγητή. Υπέρ. Yes, it looks everybody. Except, yes, okay. Uh, no? Against. Against. So we have one no vote. Uh, λοιπόν, μία αρνητική ψήφος. 116, 2, τροπολογία 2 από τον εισηγητή, 4, κατά, δεν υπάρχει αποχή, 116 παράγραφος 5 ε, υπέρ κατά καμία αποχή εγκρίνεται. Κατόπιν το 116 παράγραφος 5 τροπολογία 3 από τον εισηγητή υπέρ παρακαλώ. Μισό λεπτό, έκανε λάθος η πρόεδρος. Τροπολογία 5 υπέρ Ε, τροπολογία 5 του κυρίου Ιλτσεφ. Δύο υπέρ, κατά παρακαλώ, αποχές. Η επόμενη Λαμασούρ υπέρ, κατά, ένας κατά αποχές. Τι είστε εσείς, Υπέρ, κατά, αποχή, τι είστε. Τέσσερα, εισηγητής, αποσύρθηκε. Πάμε στην εφτά. Τροπολογία Λαμασούρη, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 ή 8 του εισηγητή υπέρ κατά Καμία αποχή εγκρίνεται. Και τελική ψηφορία υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Ευχαριστώ πολύ και ε, συγχαρητήρια. Πάμε τώρα στην επόμενη έκθεση του κ. Μέστα Σμιτ. Ένα, ένα, δύο. Υπέρ. Κατά. Τροπολογία Ράντσελ. 21. Υπέρ. seven, eight, nine, ten. Ten are four. Who are against? One. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία Άντρου Νταφ και Αλεξάνδρα Τεν. Αποσύρθηκε. Και το ίδιο και με την τροπολογία 3. Τροπολογία 23. Πάολο Ραγγέλ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Okay. It's rejected. Okay. Απορρίπτεται. 24. Αποσύρθηκε. Τροπολογία 25. Παύλο Ραγγέλ. Κατά. Αποχές. Μία. 26. Εγκρίθηκε η προηγουμένη. 26. Εδώ ζητήθηκε ψηφοφορία σε τμήματα. Υπέρ για το πρώτο τμήμα.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 Λοιπόν, υπέρ. Δεν ψηφίζουμε σε τμήματα, ψηφίζουμε συνολικά. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Είκοσι εννέα. Ραγγέλ. Πριν τα είχα κάνει λάθος. Τώρα τα κατάλαβα. Ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα. Παρακαλώ. Υπέρ. Κατά αποχές. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η τέσσερα του εισηγητή αποσύρθηκε. 30, τροπολογία 30, κυρίου Γκουαλτιέρη. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όχι, λάθος έκανε λέει πρόεδρος. Απορρίπτεται. Then the next one is... Επόμενη. Η 33. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενη. 34. 34 υπέρ. Όχι, καταπίπτει. Καταπίπτει. Εγκρίθηκε η 33 κατόπιν τούτου. Καταπίπτουν οι 32 και οι 31. Ψηφίζουμε όμως για τη 34. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Επόμενη του κυρίου Γκουαλτιέρη. Υπέρ. Κατά. Και αυτή πάλι απορρίπτεται η 35. Πάμε στην 36 του κυρίου Νταφ. Υπέρ. Κατά. εγκρίνεται. Η πέντε. Αντρουντάφ Αλεξάνδρε Τάιν. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η έξι. Της κυρίας Γιαννάκου. Υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Η 7 υπέρ κατά αποχές μία αποχή εγκρίνεται. Η 37 του κυρίου Πάσκας υπέρ παρακαλώ. κατά εγκρίνεται. Η 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 38 υπέρ κατά εγκρίνεται. Α, όχι λάθος, απορρίπτεται λέει η πρόεδρος. Η οκτώ, η επόμενη της κυρίας Γιαννάκου, υπέρ. Όχι, απορρίφθηκε, έκανα λάθος λέει η πρόεδρος. Απορρίφθηκε. Κατόπιν η οκτώ, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και η 11 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 12 των ε, Ντάφ και Αλεξανδρετάνη υπέρ κατά αποχές, άρα απορρίπτεται. Η 1 και η 13, οι τροπολογίες αποσύρθηκε και η 10 της ε, κυρία Στάιν. Πάμε λοιπόν στην 17 του Πάολο και πάλι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. <coughs> Η 14 υπέρ κατά αποχές. Πάμε στην 15 Τον Νταφ και Τάιν υπέρ κατά η 16 του Πάολο υπέρ. Κατά. Οι δύο του εισηγητή αποσύρθηκε η 18 υπέρ κατά Η 19 παρακαλώ υπέρ, κατά, η 39 Τώρα ψηφίζουμε για την 20 παρακαλώ, υπέρ. Όχι, ε, Ψηφίζουμε και πάλι για την 39. Κατά. Αποχές. Τώρα ψηφίζουμε για την 20. Υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. Καμία αποχή. Και η 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε στο, για το σύνολο υπέρ κατά εποχές, δύο εποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν για την πολύ καλή δουλειά που κάνατε και όσον αφορά το άρθρο 117 παράγραφο C, ο πρόεδρος μας δεν είναι εδώ και μίλησα και με τον σκιώδη συγητή. Κατόπιν τούτου ε, προτείνω ε, το θέμα πράγματι να τοποθετηθεί, να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη επόμενη επόμενης φοράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, καλή δουλειά, καλή σας μέρα και ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Γεια σας. Um, uh, uh, what happened to the, uh, is that the other matter?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 Χρειάζονται λοιπόν περαιτέρω διαβουλεύσει, όπως σα είπα για το σημείο αυτό. Γι' αυτό θα έλεγα να το περάσουμε στην επόμενη φορά για να έχετε κι εσεί χρόνο ελεύθερο.